αυτά τα διμερεί ζητήματα γιατί ακριβώ η κάθε περίπτωση έχει τις δικές της Αυτό το, το συνοριακό εδαφικό ζήτημα Κροατία-Σλοβενία και αυτό ήταν διμερέ. Ε, λύθηκε, ήταν ένα κράτο μέλο και κάποια τρίτη χώρα και οδήγησε στην εμπλοκή των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση τη ε, Κροατία από την άλλη μεριά. Όσον αφορά την Κύπρο, οι αποφάσει που καλούν στην υλοποίηση του πρωτοκόλλου τη Άγκυρα ήταν αποφάσει ομόφωνε μέρου τη Ένωση από του 27 όχι 25 το Σεπτέμβριο του 2005 ε, Πρόκειτο περί προπόθεση έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Είναι ευρωπαϊκό θέμα και όχι διμερέ αυτό. Και θα γίνουν, τι να σα πω, καλώ ήρθατε στο Κοινοβούλιο Και αισθάνομαι σαν έμεσα συνέντευξη τύπου και με ρωτήσατε κάτι για την κατάρριξη τη θεώρηση διαβατήριων. Είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτησή σα και σα διευκρινίζω ότι ναι, η Βοσνία Ζεγοβίνη θα έχει την ελευθερία ε, του ταξιδίου κάποια στιγμή όταν πληρούνται όλε τι προποθέσει που έχει τάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκδοση των βιομετρικών διαβατηρίων τον Οκτώβριο αρχίζει, άρχισε. Όταν δε εμεί ε, κάναμε τη σύστασή μα τον Ιούλιο δεν υπήρχε ούτε ένα σε κυκλοφορία. Τώρα η χώρα επιτάχυνε τι προετοιμασίε τη. Ήταν αυτό βασικό κίνητρο. Ούτω ώστε να τεθούν σε ισχύ κάποιοι ε, νόμοι όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια, όσον αφορά του ελέγχου των συνοριακού, όσον αφορά τα βιομετρικά διαβατήρια και κάποια άλλα σημαντικά ζητήματα, ούτω ώστε να ε, τεθούν σε ισχύ σχετικοί νόμοι και κανονισμοί τη ε, ΕΟΚ. Ήδη έγιναν συνομιλίε την περασμένη εβδομάδα για την επιτάχυνση των, της άρσης των περιορισμών ταξιδίων. Το χρειάζεται αυτό η χώρα. Χρειάζεται να, να, να, να έχει τον αναγκαίο μηχανισμό που μπορεί να το κάνει και τότε θα πληρεί τις προποθέσεις και τότε θα υπάρχει ελεύθερο ταξίδι. Ε, συμφωνώ μαζί σας, είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η χώρα υπέφερε πάρα πολλά στα δεκαετία του 90 και επομένως θα πρέπει να πάει μπροστά και να υπάρχει αυθεντικό εξευρωπαϊσμό τη κοινωνία αυτή. Οπότε, στα πλαίσια αυτά είναι σημαντική η άρση των περιορισμών 62. Ευχαριστώ. Η παρέμβασή σα ήταν πολύ χρήσιμη και πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, είχαμε ένα πραγματικό διάλογο. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής στο Στρασβούργο θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου. 6.30 ε, με 7 και 4 το απόγευμα. 6.30 με 7 και 4. Arvoisat kollegat, Καλώς ήλθατε. Καθίστε παρακαλώ. Καλώς, καλώς. Θα αρχίσουμε λοιπόν τώρα την συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με κάποια καθυστέρηση βέβαια δυστυχώς αλλά αυτό οφείλεται μόνο στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που διεξήγαγε η προηγούμενη Επιτροπή εδώ με τον ε, κύριο ε, Ρεν, τον Επίτροπο. Και ξεπέρασε το χρόνο της. Ε, τώρα μπορούμε να εξετάσουμε την ημερήσια διάταξη όπου υπάρχει μια σημαντική αλλαγή γιατί στο 4 το 4 αναγκαστήκαμε να το καταργήσουμε θέλαμε να ακούσουμε, να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον κύριο Βαν Μέβεν, αλλά δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό, διότι χρειάστηκε να μεταβεί στη Γενέβη απρόβλεπτα για να συζητήσει εκεί την έκθεση Goldstone Πάντως η γραμματεία μας κάνει την προσπάθεια να επιτύχει άλλη ε, συνάντηση μαζί του, ή δυνατόν τον Νοέμβριο. Υπάρχει ακόμη ε, διαφωνία σχετικά με την συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην έκθεση Goldstone και θα συζητήσει αυτά καθώς και άλλα θέματα όπως Μιανμάρ, Σουδάν σε πολλά από αυτά τα θέματα έχουν βρει απήχηση οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ότι ο κύριος Βαν Μέβεν θα προσκληθεί και στην Επιτροπή Εξωτερικών για να ε, ακουστούν και εκεί οι απόψεις του για την έκθεση Goldstone. Επιθυμώ επίσης να πω ότι Είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Επίτροπο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών δηλαδή, που θα είναι στις Βρυξέλλες σύντομα, γιατί τα Ηνωμένα Έθνη ανοίγουν εδώ γραφείο στις Βρυξέλλες τώρα και θα είναι χρήσιμο να μπορέσουμε να συναντηθούμε με τον κύριο Λόχ Μπίλερ τον κύριο Χάουιτ, την κυρία Αντρικένε. Είμαι βεβαία ότι πρόκειται να συνεργαστούν πολύ με τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει και δικό της έργο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δίνοντας έτσι το καλό παράδειγμα. Εξάλλου, προβλέπεται και επίσκεψη μέλους της γερουσίας της Νιγηρίας που βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την ώρα συνοδεύοντας τον προεδρεύοντα δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και σε μια συνάντηση με μια οργάνωση που λέγεται Βουλευτές Υπερασπιστές των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις του γερουσιαστού αυτού. Μπορείτε λοιπόν να συμφωνήσετε με την ημερήσια διάταξη. Καλώς. Έγινε λοιπόν και αυτό και μένει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 10 η Σεπτεμβρίου. Τα εγκρίνεται, έχει καλώς. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Ο πρόεδρος μας κύριος Μπούσεκ στις 10 Οκτωβρίου οργάνωσε την ημερίδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε στην ομιλία του ότι για την ώρα η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, όχι της Ένωσης, η οποία εξακολουθεί να εφαρμόζει την ποινή του θανάτου είναι η Λευκορωσία. Είναι εξάλλου σημαντική και η επέτειος της 20 ετίας από την υπογραφή της Συμφωνίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Είναι γνωστό βέβαια δυστυχώ ότι σε ορισμένε χώρε εξακολουθούν και εκτελούν θανατικέ ποινέ σε βάρο και ανηλίκων. Στο Ιράν την Κυριακή εκτελέστηκε ένα ανήλικο που λεγόταν Μπεχτούν Σετζάι και πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταματήσει αυτό. Στην Κίνα εξάλλου μάθαμε ότι καταδικάστηκαν σε θάνατο έξι Ουιγκούρ μετά από τις ταραχές που σημειώθηκαν τελευταία στο Ουρούμτσι. Οι χώρες μέλη ζήτησαν να μπορέσουν να αποστείλουν παρατηρητές στις σχετικές δίκες αλλά οι Κινέζοι ούτε καν ανακοίνωσαν πού διεξάγονται οι δίκες. Έχουμε τώρα επίσης μια σημαντική έκθεση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε επεξεργασία σχετικά με την εξωτερική υπηρεσία που θα εξαρτηθεί βέβαια από την θέση εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Μας έχει ζητηθεί να συντάξουμε γνωμοδότηση για το θέμα. και να το συζητήσει η υποεπιτροπή μας. Εμείς έχουμε ορισμένες τροπολογίες της κυρίας Λόχπιλ και δικές μου για να μπορέσουμε να περιλάβουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις πτυχές των εξωτερικών μας σχέσεων. Ας είμαστε λοιπόν όλοι οι παρόντες και παρούσες για να ψηφίσουμε υπέρ της τροπολογίας αυτής. Τώρα, άλλο θέμα είναι η δημοκρατική συνένεση. για τα οποία έχουμε υποβάλει ορισμένες, ε, προτα... ορισμένες ερωτήσεις για την ε, Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ώστε να γραφτούν στην ημερήσια διάταξη της μήνυ Ολομέλειας του Νοεμβρίου. Είναι σημαντικό το χρονικό αυτό σημείο διότι θα μας επιτρέψει να επηρεάσουμε τις συζητήσεις που θα γίνουν μετά στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Η Γραμματεία συντάσσει πρόταση ψηφίσματος που θα αποτελέσει τη βάση Δεν ξέρουμε βέβαια πότε ακόμα θα γίνει η συζήτηση αυτή. Το τελευταίο που θέλω να θέσω υπόψη σας είναι σχετικά με το Ουσμπεκιστάν. Οι Υπουργοί Εξωτερικών προτίθεται να συζητήσουν την απαγόρευση χρήσεως όπλων στο Ουσμπεκιστάν στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Υπάρχει και ε, το ενδεχόμενο να συζητηθούν κυρώσεις, επιβολή κυρώσεων. Κυρώσεις που επιβάλλονται ήδη στο Σμπικιστάν από το 2005. Λόγω του ότι τότε είχαν σημειωθεί πολύ φόνοι στην πόλη Αντιτζάν. Αναμένουμε ε, και μια διεθνή έκθεση για τα θέματα αυτά, για τα γεγονότα μάλλον εκείνα, της Αντιτζάν. Οι αρχές του Ουσμπεκιστάν δυστυχώς δεν έχουν επιτρέψει ε, τη διεξαγωγή ιασδήποτε έρευνας. Και γι' αυτό εμείς ζητούμε τώρα να επιβληθεί, επιβλήθηκε μάλλον ήδη απαγόρευση έκδοσης προξενικών θεωρήσεων βίζα από τον περασμένο Οκτώβριο. Δυστυχώς το Συμβούλιο δεν ασχολήθηκε με τα γεγονότα του Αμπιτζάν. Θεώρησε το Συμβούλιο ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα στο Σμπεκιστάν τώρα και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ενώ εμείς γνωρίζουμε ότι η κατάσταση του Ζουμπικιστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα προκαλεί μεγάλες ανησυχίες. Ένα από τα προβλήματα είναι η παιδική εργασία εκεί. Ώστε σας παρακαλώ παρακολουθήστε προσεκτικά την εξέλιξη του θέματος για να μπορούμε να συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής. Ίσως μπορούμε να αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση. Κυρία Λόχπιλ πρώτη. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Στις 26 και 27 Οκτωβρίου οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών θα αποφασίσουν εάν θα άρουν το εμπάργο όπλων που βαραίνει το Ουσμπεκιστάν. Αυτό θα εμποδίσει οποιασδήποτε ε, έρευνες για την σφαγή στο Αντιτζάν. Το θέμα είναι τι σημαίνει αυτό για τις οικογένειες και για τα θύματα. Και επιπλέον θα είναι και ένα κόλαφος για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουσμπεκιστάν το να στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τέτοιο μήνυμα ότι δηλαδή δεν παίρνει πολύ στα σοβαρά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί. Επομένως θα πρέπει να θέσουμε αυτό το ερώτημα στη γερμανική κυβέρνηση, γιατί βλέπουμε ότι διστάζει να ψηφίσει για τη διατήρηση του εμπάργου όπλων. Αν γίνεται λοιπόν, θα ήθελα η Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος να στείλει μια επιστολή στον κύριο Μπίλτ και να δείξουμε στεναρότητα. Να πούμε ότι στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπάρχει ουσιαστική βελτίωση, ότι έχουν ε, ε, γίνει συζητήσεις για την, ε, τις φαγές του Αντιτζάν, αλλά σε καμία περίπτωση αυτές οι έρευνες δεν είναι αμερόληπτες, ανεξάρτητες και ευρείες, πλήρεις. Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κυρία Λοχμπίλερ. Κύριε Όουιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο γενικά σχόλια για τις ανακοινώσεις σας που δεν σχετίζονται με το θέμα του Ουσμπεκιστάν. Καταρχάς, καλωσορίζω το γεγονός ότι ρυθμίσαμε τα θέματα με την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων και δεν υπάρχουν επικαλύψεις των συνεδριάσεών μας, γιατί συνέβαινε αυτό στο παρελθόν και αυτό ήταν πάρα πολύ κακό. Ε, μερικές φορές πρέπει και εμείς λοιπόν να επιμένουμε, να επιμείνουμε στο ότι έχει η πρωτοκαθεδρία η δική μας ατζέντα. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν επικαλύψεις των συνεδριάσεων, να μην γίνουν την ίδια ώρα. Δεύτερον, ε, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά από ό,τι ξέρω ο εκδημοκρατισμός θα συζητηθεί την Τρίτη ε, στο Στρασβούργο. Ε, ίσως έχετε πιο φρέσκες πληροφορίες. Ίσως ε, ληφθεί απόφαση σήμερα το απόγευμα. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να συνεργαστούμε για το ψήφισμα. Αν όμως συζητηθεί όντως την Τρίτη στο Στρασβούργο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ, κύριε Χάουιτ. Από ό,τι ξέρω, οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων θα αποφασίσουν σήμερα για να δούμε εάν το θέμα του εκδημοκρατισμού θα συζητηθεί τελικά στην Ολομέλεια ή όχι. Πάντως θα ήταν καλό νέο να γίνει την επόμενη εβδομάδα την η συζήτηση αυτή. Θα μπορούσαμε ίσως να ζητήσουμε από τους γενικού Γραμματεί να περάσουν το μήνυμα α, στους πρόεδρους των πολιτικών ομάδων. Για το Ουσμπεκιστάν, θέλετε το λόγο. Ναι, πράγματι κυρία Πρόεδρε, για το Ουσμπεκιστάν. Από εδώ και μία δεκαετία είμαι μέλος της αντιπροσωπείας για τη σχέση με το Ουσμπεκιστάν. Εδώ και ένα χρόνο δεν μπόρεσα βέβαια να επισκεφθώ τη χώρα αυτή. Θέλω να επισημάνω ωστόσο το εξή. Σε όσα κάνουμε θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις πρόοδους που όντως επιτελεί η χώρα αυτή. Όποιος γνωρίζει την ε, εκπρόσωπο έχει την εντύπωση, αποκομίζει αμέσως την εντύπωση ότι θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να την ενισχύσουμε. σχετικά με τις θανατικές εκτελέσεις. Μιλήσατε πριν για θανατικές εκτελέσεις ε, νέων ανηλίκων. Το Ουσμπεκιστάν κατήργησε τη θανατική ποινή. Να λοιπόν μια πρόοδος. Είναι μικρή, ίσως πρόκειται για ε, μια πορεία που γίνεται ούτε καν σε εκατοστά αλλά σε χιλιοστά αλλά ωστόσο υπάρχουν άλλες χώρες που δεν κάνουν ούτε αυτή την πρόοδο χιλιοστών. Θα έλεγα λοιπόν να έχουμε πάντοτε μια ε, σαφή αίσθηση των, των πραγματικών διαστάσεων των προβλημάτων και των προόδων. Ευχαριστώ κυρία Γέγκλερ. Ε, επανέρχομαι σε αυτά που είπε η κυρία Λόχ Μπίλερ. Ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μαζί με τον Αντιπρόεδρο να έρθει ο κύριος Μπίλτα στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα. Ίσως ε, η κυρία Γέγγελ, η κυρία Μπίλερ ε, θα μπορούσαμε θα μπορούσαν να είναι παρούσες ε, σε αυτή τη συνεδρίαση, εφόσον τις ενδιαφέρει. Για να δούμε τι θα γίνει με την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι σε αυτές τις χώρες. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Αυτό και θα κάνουμε. Μαζί με τον Αντιπρόεδρο θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε αυτή τη συνάντηση. Ωραία. Και τώρα πάμε στο κυρίω πιάτο. Έχουμε, και θα έχουμε μάλιστα και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, μια και δεν θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Άλεξ Βαν Μεύεν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λοιπόν, πρόκειται για την χρηματοδοτική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα θέμα το οποίο ε, μου αρέσει όλος ιδιαίτερος. Ε, θα υπάρξει μια ενδιάμεση έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μας παρουσιαστεί για το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι αυτή η ενδιάμεση έκθεση είναι μια συνήθις έκθεση που παρουσιάζει η Κομισιόν και αφορά τα πάντα, το χρηματοδοτικό, ό,τι έχει να κάνει με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Επίσης θα έρθει και ο Γενικός Διευθυντής, ε, ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, εν συνεχεία, ο Λέωνορ Μπασάν, που είναι και εδώ, στην αίθουσα, και η συντονίστρια για το δίκτυο Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ένα δίκτυο το οποίο εξέτασε το χρηματοδοτικό αυτό μέσο. Έχουμε και την Αλεξάνδρα Μανκάροφ ε, της οργάνωσης Κονκόρντια. Πρόκειται, εκπροσωπεί ένα δίκτυο συνεργασίας πάλι η κυρία αυτή. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τα άτομα αυτά για τη σχέση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ακούσουμε καταρχήν τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να μας πείτε σας παρακαλώ, ε, περί τίνος πρόκειται, τι είδους χρηματοδοτικό μέσο είναι αυτό. Θα θέλαμε τι, να μας πείτε τι πετύχαμε χάρη σε αυτό το χρηματοδοτικό μέσο. Εν συνεχεία, θα πάρουν το λόγο οι υπόλοιποι ομιλητές για να μιλήσουν για τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στρατηγικούς τρόχους που θα υλοποιήσει αυτό το μέσο μέχρι το 2013. Εν συνεχεία θα ακούσουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ο εκπρόσωπος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην εισαγωγή σας είπατε ότι η Ευρώπη και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να είναι παρόντα και να έχουν μια μεγάλη ορατότητα. Θα προσπαθήσω να το αποδείξω αυτό. Από το 2006 έχουμε αυτό το ευρωπαϊκό, αυτό το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι διάδοχος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και είναι το χρηματοδοτικό μέσο υπό το οποίο η κοινότητα δίνει βοήθεια ανά τον κόσμο για την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Μιλάμε τώρα για χρηματοδότηση τρίτων χωρών. Το μέσο αυτό προοικοδοτείται με 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007 και μέχρι 2013. Εάν δεχθούμε να πάνε αποστολές ε, εκλογικής παρατήρησης τότε θα πρέπει να καταβληθούν 115 ε, εκατομμύρια σε αυτές τις αποστολές. Το μέσο αυτό συνεισφέρει στην ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών παντού σε όλο τον κόσμο. Η χρηματοδότηση υπό αυτό το μέσο είναι συμπληρωματική με την κοινοτική βοήθεια που χορηγείται μέσω της διμερούς συνεργασίας η βασική δύναμη αυτού του μέσου έγκυται στην ικανότητά του να λειτουργεί ανεξάρτητα, χωρίς τη συνένεση των κυβερνήσεων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να εστιάσουμε σε ευαίσθητα πολιτικά θέματα, στη συνεργασία με την τοπική κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις της, που χρειάζεται να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους από τις δημόσιες αρχές. Το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ακριβώς για αυτό το λόγο, μπορεί να, παίξει ρόλο σε χώρες που θα μπορούσαμε να τις περιγράψουμε ως δύσκολες, δύσκολους εταίρους και όπου οι θεμελιώδεις ελευθερίες κινδυνεύουν και όπου Μπορεί να υπάρχουν και γεωγραφικά προβλήματα. Το μέσο ε, λειτουργεί μέσω διαγωνισμών ή στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με διεθνείς οργανώσεις για να προωθήσουμε την οικοδόμηση της δημοκρατίας, το να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως το κράτος δικαίου, την ε, διεθνή δικαιοσύνη και την προώθηση των θεμελιωδών ελευθεριών μεταξύ άλλων. Μέχρι στιγμής πάνω από 100 προτάσεις έχουν υποβληθεί από διάφορες αντιπροσωπείες, προτάσεις υποβολής ενδια... Ε, προκήρυξης ενδιαφέροντος, ε, κάτι που μεταφράζεται σε 400 προγράμματα παγκοσμίως. Από αυτά τα 400, πάνω από 300 είναι τοπικά προγράμματα της τοπικής κοινωνίας των πολιτών σε 70 διαφορετικές χώρες. Προγράμματα τα οποία τα διαχειρίζονται απευθείας οι αντιπροσωπείες της κοινότητας επιτόπου. Τα υπόλοιπα είναι διεθνή προγράμματα ε, που αφορούν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες σε χώρες και περιοχές όπου κινδυνεύουν τα μάλα. Εκεί έχουμε 27 προγράμματα που είναι εξελίξη και 19 που είναι σε φάση ετοιμασίας. Η καταπολέμηση της ε, θανατικής ποινή. Εκεί για αυτήν έχουμε 8 προγράμματα και 5 εντογενάστε. το ε, προγράμματα για το βασανιστήριο. Έχουμε 7 που τα διαχειριζόμαστε από εδώ από τις Βρυξέλλες και 25 από τις αντιπροσωπείες μας ανά τον κόσμο και τέλος για τους υπερασπιστές των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 11 μεγάλα προγράμματα με μηχανισμούς ε, υποστήριξης και δυνατότητα ε, νέας χορήγησης δανείων και κονδυλίων και βεβαίως έχουμε πέντε προγράμματα για την υποστήριξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Το 2009 και 2010 οι αιτήσει συνέχισαν να σειραίουν. Οι από το, πλαίσιο, το διαρκές πλαίσιο προκήρυξης προσφορών και αφορούν χώρες και περιοχές που, όπου κινδυνεύουν η δημοκρατία και τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Ε, επίσης, τέτοιες προτάσεις για, το, για να καταπολεμήσουμε τα πασανιστήρια ε, οι προθεσμίες αυτές κλείνουν σήμερα. Επίσης, Τρεις, άλλοι διαγωνισμοί ε, θα ξεκινήσουν επόμενο μήνα. Καταρχάς, μία, για να υπάρχει αποτελεσματική λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ε, θα κλείσει προθεσμία στο τέλος Οκτωβρίου. Ένα, για διπλώματα μάστερ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εκδημοκρατισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ξεκινήσουν ε, οι προσφορές το Δεκέμβριο και δράσεις υπό για την υποστήριξη των ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα ξεκινήσουν οι προτάσεις να υποβάλλονται το πρώτο εξάμεινο του 2010. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύψουμε την περίοδο 2007-2010 μέχρι τον Ιούνιο του επομένου έτους. Το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επίσης λειτουργεί μέσω των ε, στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με διεθνείς οργανώσεις για να προωθηθεί η οικοδόμηση της δημοκρατίας, να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως το κράτο δικαίου, η διεθνής δικαιοσύνη, το διεθνές δίκαιο και η προώθηση των θεμελιώδων ελευθεριών. Αυτά μεταφράζονται σε περίπου 20 στοχευμένες δράσεις με στρατηγικούς εταίρους που συμπεριλαμβάνουν το Ηνωμένα Έθνη και το Γραφείο του ΙΠΑ του Εκπροσώπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Συμβούλιο της Ευρώπης ή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το μέσο επίσης υποστηρίζει ε, διπλώματα μάστερ για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, με προγράμματα συνεργασίας ΟΗΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλες ερευνητικές δραστηριότητες ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προωθούν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Αυτό σημαίνει δύο υποτροφίες, υποτροφίες για τα διπλώματα αυτά μάστερ. Επίσης, ε, υποστήριζουμε τα Βαλκάνια, την Λατινική Αμερική, την Νότια Αφρική και την Ασία και τον Ειρηνικό. Ε, οι αποστολές ε, παρατήρησης των εκλογών επίσης χρηματοδοτούνται υπό αυτό το μέσο. Αποτελούν ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Είναι ένα από τα λίγα ολοκληρωμένα μέσα για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επικεφαλής της αποστολής ε, διορίζεται από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή ε, Ανάπτυξης και οι παρατηρητές προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Οι αποστολές αυτές οργανώνονται από και την χάνουν διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ε, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο υποστηρίζουμε διάφορα προγράμματα. Ε, τα περισσότερα κονδύλια περνάνε μέσω του ε, μέσου καλής γειτονίας. Συνήθως προωθούμε τα πιο μικρά προγράμματα που αφορούν συγκεκριμένες χώρες ε, με σκοπό να βελτιώσουμε την πρόσβαση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών των ε, ενδιαφερόμενων χωρών. Η διαχείριση των ε, προγραμμάτων αναχώρα γίνεται από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 77 χώρες έχουν λάβει κονδύλια το 2009 και αυτό το νούμερο θα αυξηθεί σε 92 χώρες το 2010. Οι αντιπροσωπείες εκλογικής παρατήρησης ε, συνεχίζονται στο Αφγανιστόν, τη Βολιβία, τη Μοζαμβίκη και την ακτή του Ελεφαντοστού. Και αυτό αφορά τους τρεις τελευταίους μήνες του 2009. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Τώρα, ο κύριος ε, Ρολφ Τίμανς ε, παρίσταται από την ε, Υπηρεσία Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μου ζητήσατε να σας μιλήσω για το νέο πλαίσιο που θα έχουμε για την πολιτική μέσα του 2013 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρόκειται για υποχρέωση που αναλάβαμε ε, να γίνει 2009-2010 ε, μια αναθεώρηση κάθε ενίσχυσης χρηματικής περιλαμβανομένων και της υπάτης αρμαστίας και επίσης να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια αναθεώρηση της στρατηγικής του 2007 τον Αύγουστο. Όσο αφορά την υπατηρομοστία, εμείς πιστεύουμε ότι η περίοδος εφαρμογής ουσιαστικά αυτής της στρατηγικής είναι πάρα πολύ σύντομη τόσο ώστε να μπορέσουμε να επιφέρουμε κάποιες ουσιώδεις μεταβολές. Το ιστορικό πλαίσιο ξέρετε ποιο είναι ότι μόλις τον Αύγουστο του 2007 ε, υιοθετήθηκε αυτό και η ουσιαστική εφαρμογή άρχισε το δεύτερο εμείς του 2008 ε, τότε έγιναν οι προδιαγωνισμοί κλπ. Ούτε έτρεξε τίποτα άλλο εκτός από αυτές τις αποστολές παρατήρησης εκλογών και ούτω ώστε δεν έχουμε κάποιο είδου ε, κριτήρια, κάποιο είδου ιδέε για την αποτελεσματικότητα τη στρατηγικής του 2007. Επίσης, στα πλαίσια ε, αυτών των, των, των προετοιμασιών της αναθεώρησης Έχουμε απευθυνθεί σε κάποιε εταιρείε συμβούλων, τόσο ώστε να δουν επί τόπου πώ έχουν τα πράγματα και όπω ακούσατε, έχουμε μια σειρά χωρών ε, που μα απασχολούν και ε, στι περισσότερε από αυτέ τι ε, δουλειέ το ώστε που έχουμε ανοίξει. Έχουμε ένα feedback από αυτού του ε, συμβούλου, ούτω ώστε ε, ε, δεν θα πρέπει να βιαστούμε, μην κάνουμε πάρα πολύ νωρί την αναθεώρηση. Ταυτόχρονα δε οι εταιρείε συμβούλων μα είπαν ότι θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε αυτέ τι πέντε στόχου κλειδιά ότι θα πρέπει και στην επόμενη περίοδο 10 έως 13 να συνεχιστούν όπως και στην απόφαση του 2007. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι οι μεταβολές τις οποίες θα επιφέρουμε ή θα προτείνουμε να γίνουν σε αυτή την στρατηγική, στα πλαίσια της τα θα είναι περιορισμένες επί της ουσίας. Οι στόχοι κλειδιά θα παραμείνουν και θα εισαγάγουμε κάποιες πινελιές σε διάφορα σημεία Ήδη άρχισαν οι συναντήσεις με την ΟΚΕ και την Επιτροπή των Περιφερειών, με οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, από όλο το φάσμα των, των εμπλεκομένων σε υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει και μια συγκεκριμένη μνήμα που θα διατυπώσει στο μέλλον όσον αφορά τη στρατηγική που χρειάζεται για να υποστηρίξουμε τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα πέραν των ε, ε, πολιτικών δικαιωμάτων. Επίσης, ε, θα τονίσουμε την σημασία του διαλόγου, ούτως ώστε να προαχθεί η ειρήνη αλλά και η πρόληψη των κρίσεων. Μπορείτε να δείτε επομένω διάφορα στοιχεία τα οποία θα χαρακτηρίσουν τι προτάσει μα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα όσα μας είπαν οι σύμβουλοι. Ε, όμως υπάρχουν κάποιες ε, ουσιαστικές αλλαγές ε, στην αναθεωρημένη μελλοντική στρατηγική. Αυτό θα αφορά την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που προβλέπονται. Αυτό σημαίνει ότι επειδή θα αυξηθεί η ζήτηση της κοινωνίας των πολιτών στις τρίτες χώρες σε σχέση με το ότι ισχύει σήμερα θα αυξήσουμε ελαφρώς το ποσοστό των επιχειρήσεων αναχώρα. Και όσο με τι περιφερειακές ε, επιχειρήσεις ε, θα υπάρξει μια μικρή συγγνώση γιατί μέχρι τώρα τα πράγματα δεν πήγανε προς ποιότητος των επιχειρήσεων όπως θα θέλαμε. Επίσης, η στρατηγική μας θα καλύψει την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κατά των ανηλίκων, που είναι καθημερινές γραμμές που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό έχει ξεκινήσει το 2007, αλλά θα προσθεθεί και τώρα και τις σχετικές ποσοστώσεις ε, που ίσχυαν θα τις ε, πάυσουμε και θα γίνει αλλιώς η σχετική χρηματοδότηση. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι θα είναι περιορισμένες οι μεταβολές στην στρατηγική μας στο μέλλον. Ελπίζουμε δε ότι με μια τέτοια προσέγγιση θα πάρουν το πράσινο φως από τα κράτη-μέλη αλλά και από τη Διαχειριστική Επιτροπή της, της Αρμοστίας αλλά ότι βέβαια και εσείς θα συνενέσετε. Ο πλευράς χρονοδιαγράμματος, εν τέλει, πρέπει να σας πω ότι η αναθεωρημένη στρατηγική θα υποβληθεί στην Διαχειριστική Επιτροπή της Πατσαρμοστίας 14 και 15 Δεκεμβρίου. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι αμέσως όλοι μαζί θα εγκριθεί, αλλά στη συνέχεια θα σας διαβιβαστεί το έγγραφο για να κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θα υπάρξει επίσης άλλο ένας γύρος εννοήσεων με την κοινωνία των πολιτών. Δεύτερο γύρος μετά τα όσα προηγήθηκαν τον Ιούλιο και ελπίζουμε ότι θα τηρηθεί η προθεσμία που έχει τάξει για όλε τι αδικίε η Κομισιόν τέλος Μαρτίου του 2010 δηλαδή σε αυτό το χρονικό πλαίσιο κινούμεθα. Τελευταία μου παρατήρηση, Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε. Δεν πρόκειται μόνο για αναθεώρηση ε, στρατηγικών, πρόκειται και για αναθεώρηση των κανονισμών που διέπουν τις σηματοδοτικές ενέργειες. Και όσον αφορά τον κανονισμό της υπερσαρμοστίας της 28 Δεκάτου 2006, πολύ ελάσσονες προσαρμογές θα γίνουν για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα του ΦΠΑ όσον αφορά την εξωτερική βοήθεια. Καμία ουσιαστική θα γίνει, αλλαγή δεν πρόκειται να γίνει, τουλάχιστον να προτείνουμε εμεί. Επομένω, η Επιτροπή σα θα ενημερωθεί, θα λάβει την συνολική πρότασή μας όπου θα για αυτό το θέμα του ΦΠΑ. Και θα καλύψουμε και τα όσα τάσει το, το, το, μέσο της αναπτυξιακής βοήθειας. Κύριε Τίμαν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει Πρόεδρος. Ακούσαμε τον κύριο και αλλά και τον κύριο Τίμαν, ακούσαμε μένω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα δώσουμε το λόγο στι μη κυβερνητικέ οργανώσει που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτή τη ε, προσπάθεια αλλά βέβαια είναι και χρήστες κατά κάποιο τρόπο του συστήματος. Η κυρία Ρεμπάς επίσης έχει συντάξει κάποιο έγγραφο όσον αφορά το δίκτυο των οργανώσεων για τον εκδημοκρατισμό. Σας ευχαριστώ. Θα αρχίσω εγώ, μετά η φίλη μου Λεωνόρα Λέγομαι Αλεξάνδρα Μακπρόφ και είμαι της Plan International από τις πιο μεγάλες ε, οργανώσεις για την ανάπτυξη των παιδιών και που ανήκουμε στην οικογένεια της Concord και μιλώ ως ενεργό μέλος της Concord. Η Concord, εφόσον δεν τη γνωρίζετε ορισμένη, είναι μια ε, ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Ενώσεων με πάνω από 1.600 οργανώσεις στις 27 χώρες μέλη μέσω δικτύων εθνικών πλατφόρμων που εκπροσωπούν χιλιάδες Ευρωπαίων πολιτών. Χαιρόμαστε για την ευκαιρία που μας δίνει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να εκφράσουμε την άποψή μας, ε, άποψη των μη κρατικών οργανώσεων ανάπτυξης Νομίζουμε ότι πρόκειται για ένα βήμα προ τα εμπρό, προ την κατεύθυνση ενό πιο επικοδομητικού στρατηγικού διαλόγου με τα τρία θεσμικά όργανα. Είμαστε σε διαρκή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της EuropeAid, αλλά είναι σημαντικό να αναπτύξουμε διάλογο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, το οποίο εποπτεύει του σχετικού μηχανισμού, όχι μόνο με την ε, Επιτροπή Ανάπτυξης, αλλά και με τη δική σας υποεπιτροπή, διότι βρίσκουμε ότι οι δύο αυτές επιτροπές είναι συμπληρωματικές. Επειδή λοιπόν είσαστε συμπληρωματικέ, θεωρώ η Concord και η δική μας ε, ε, οργάνωση είναι επίσης συμπληρωματικέ. Έχουμε τη δική μας, έχουμε και τη Λεωνόρ που είναι των παιδιών και έχουμε κοινού ε, στόχους για θέματα ανάπτυξης, καταπολέμησης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού κλπ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανάπτυξη είναι στην ουσία δύο Πλευρέ του ίδιου νομίσματος, δύο όψει του ίδιου νομίσματος. Τελευταία έχουμε αναλάβει την, έχουμε ε, αντιμετωπίσει την πρόκληση του λεγόμενου mainstream, δηλαδή να περάσουν σε όλες τις πτυχέ της ζωής ε, τα θέματα που μας απασχολούν και είναι σημαντικό οι στόχοι των οργανώσεών μας ε, να θεωρηθούν συμπληρωματικοί και να τους δοθούν οι ίδιες προτεραιότητες μέσα στα πλαίσια του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφωνούμε όλοι ότι η προσέγγιση βασισμένη ανθρώπινα δικαιώματα ε, μπορώ να σας δώσω ορισμένες σύντομες συστάσεις και σχόλια για τον ίδιο το μηχανισμό. Η Concord έχει εντοπίσει τρία βασικά θέματα που θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας. Πρώτο, η διαδικασία διαβούλευσης. Αναγνωρίζουμε ότι η συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην διαδικασία είναι πλέον συνεκτικότερη από ε, παλαιότερα και κυρίως στο επίπεδο των ε, αρχηγείων μας εδώ στις Βρυξέλλες. και νομίζουμε ότι ακόμα δεν είναι επαρκής η ε, διαβούλευση και δεν υπάρχει επαρκής πίεση στις αντιπροσωπείες για να διαβουλεύονται. Μία σύντομη ανάλυση της Concord στα μέλη της και έκλεισε το μικρόφωνο της ε, κυρίας. Ε, λάβαμε απαντήσεις από τα μέλη μας που δείχνουν ότι σχεδόν καθόλου διαβούλευση δεν έχει γίνει στο τοπικό επίπεδο και εγώ με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης έχω έρθει σε επαφή με τα γραφεία μας και εκτός από την Ουγγάντα και Ρουάντα δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση για την σύνταξη του ε, σχεδίου του ε, επομένου χρόνου. Δεν λέω ότι δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση. Πάντω τα γραφεία μας δεν έχουν καμία σχετική πληροφορία. Ίσως ακούγεται το ύφος μου, μου λίγο προκλητικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με τις τοπικές ε, οργανώσεις. Δεν είναι δυνατόν να τους υπαγορεύουμε εμεί ποιε είναι οι ανάγκε τους. Ο προπολογισμό που είναι διαθέσιμος για την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού είναι πολύ μικρός. Είναι σχετικά περιορισμένος, λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να μπορέσουν οι μηχανισμοί αυτοί να εκπρόσουν τους σκοπούς τους, είναι απαραίτητο ο προϋπολογισμός να αυξηθεί αντίστοιχα. Όπως ε, τονίζει και το Ελεκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του, είναι ότι τα δημοσιονομικά μέσα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά με Καλή ποιότητα προτάσει, οι οποίες τελικά απορρίπτονται λόγω της έλλειψης ε, χρηματοδοτικών μέσων και αυτό είναι ιδιαίτερα ε, αληθέ για το EDIHR. Εν τέλει, πολλοί αναρωτιούνται έχει νόημα να υποβάλουμε αιτήσει για χρηματοδοτικά μέσα από τον προπολογισμό αυτό όταν υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός. Όπως άλλωστε είπε ο κύριος Τίμανς προηγουμένως, η ανακοίνωση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ορισμένες προσκλήσεις ενδιαφέροντος μπορεί να μην γίνουν ε, του χρόνου. Και τέλος, ό,τι αφορά την διαθέσιμη χρηματοδότηση, υπάρχει η τάση των διεθνών δωρητών να περάσουν σε άμεση ενίσχυση των κρατικών προπολογισμών αντί να χρηματοδοτούν οργανώσεις τη κοινωνία των πολιτών. Ενώ αυτό θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να φτάσετε στους πιο, στα πιο τροτά μέρη ε, του πληθυσμού. Τέλος, θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα βελτίωση των διαδικασιών προσκλήσεων εκδηλώσεως ενδιαφέροντο, γιατί για την ώρα δεν υπάρχει δεν υπάρχουν κανονισμοί για υπάρχουν ρυθμίσει για, αυτού, για τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος για το EIDHR. Άλλε είναι ανοιχτέ, άλλε διαδικασίε είναι κλειστέ. Και αυτά οδηγούν σε σημαντική έξτρα επένδυση και χρήματος και χρόνου χωρίς τα αποτελέσματα από πλευρά των οργανώσεων των, της κοινωνίας των πολιτών. Χάρηκα που άκουσα τον κύριο Τίμανς να λέει ότι το θέμα του φόρου προς τη θέμενη αξία ίσως επιληθεί για τις μελλοντικές προκλήσεις ενδιαφέροντος, αλλά γενικά υπάρχει σαφής έλλειψη ε, ε, ευκαμψίας και καμιά φορά οι διαδικασίες είναι δυσκίνητες και δυσανάλογες. Νομίζουμε ότι οι διαδικασίες αυτές δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικές και συμπεραίνοντας θα ήθελα να ευχαριστώ και πάλι την Επιτροπή σας που δίνει στην Κονκούρ τη δυνατότητα να ε, αναπτυχθεί. Όπως είπα προηγουμένως, είναι οι δύο ε, πλευρές του νομίσματος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των προσπαθειών μας και ιδιαίτερα η δική σας υποεπιτροπή έχει τη δυνατότητα να ε, κάνει καλύτερο συνδυασμό των προσπαθειών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Χθες ε, η οργάνωση Concord ήταν εδώ για τη δημοσίευση του εγγράφου της που αφορά διάφορους τομείς Ξέρετε πολύ καλά ότι ασχολούμαστε πολύ και συνεργαζόμαστε πολύ με την ε, Επιτροπή Ανάπτυξης για να προωθήσουμε τα αναπτυξιακά θέματα. Και θυμάμαι ότι συζήτησα με τον πρόεδρο Μπούζεκ ε, το θέμα της ε, συνεκτικότητας των όσων κάνουμε. Και μου είπε ότι καλό θα ήταν να συζητήσουμε με οριζόντιο τρόπο αυτά τα θέματα στο Κοινοβούλιο. Ίσως θα μπορούσαμε να εμπλέξουμε και την Επιτροπή Γεωργίας. Γιατί και το θέμα της επισητιστικής ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσαμε να εμπλέξουμε επίσης και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Μου ζητήθηκε λοιπόν να κάνω μία πρόταση γιατί το θέμα είναι πραγματικά οριζόντιο και μας αφορά όλους καθημερινά. Ο επόμενος ομιλητής. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, είμαι Λεωνόρ Βασάρ. Ε, δουλεύω στο Διεθνές Ίδρυμα για την Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι τμήμα ενός ατύπου δικτύου που, όπου συνεργάζονται διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, Συμμετέχουν πάνω από 40 μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο και συνεργάζονται και με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για διάφορα θέματα που αφορούν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρούμε ε, ότι το δίκτυο αυτό δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσπαθεί να εντάξει την ε, διάσταση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές εξωτερικής χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς από πλευράς μας, ως δίκτυο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, πιστεύουμε ότι είμαστε συνομιλητές και έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε ε, γιατί σας δίνουμε ουσιαστικά πληροφορίες από τους ε, εταίρους μας σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή είμαστε ένα σημάντας διαβίβασης ε, κάποιων απόψεων στα θεσμικά κοινοτικά όργανα. Ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας δίνει την δυνατότητα να μιλήσουμε εδώ στην Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ελπίζουμε ότι αυτό είναι ένα παραπέρα βήμα για τη βελτίωσμένη συνεργασία και τον ε, διάλογο μαζί σας και για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και για αυτό το ιδιαίτερο θέμα του χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα του μέσου αυτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τον, την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών από πλευράς Κομισιόν Χαιρόμαστε, η οποία είναι, χαιρόμαστε γεγονός ότι είναι διατεθειμένη να μας δώσει διάφορες πληροφορίες και να συζητήσουμε διάφορα θέματα που μας απασχολούν. Αλλά πραγματικά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν. Έχω να θέσω ένα συγκεκριμένο αίτημα, υπόδειξη, πώς να το πω. Καλό θα ήταν, χρήσιμο θα ήταν, αφού σας δώσουμε εμείς κάποιες πληροφορίες, να μας δίνετε κι εσείς κάποιες πληροφορίες από τη μεριά σας. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία εκμάθηση. Ειδικά για εμά, τι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, δεν γνωρίζουμε τις τεχνικές λεπτομέρειε χρηματοδότηση. και συχνά έχουμε την αίσθηση ότι δεν έχετε λάβει υπόψη σας τι τις προτάσεις γιατί πραγματικά είμαστε λίγο εκτό θέματο. Καλό θα ήταν λοιπόν να μα ε, απαντάνε ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, να μα δίνουν πληροφορίε και αυτά με τη σειρά του. Γιατί εμεί δίνουμε, αλλά να παίξετε κι εσεί αυτό το ρόλο. Σε ό,τι αφορά... Αυτά σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις στην Ευρώπη. Από την άλλη που και ο, Αλε... ο υπάρχει μια σημαντική διαδικασία διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο, στις διάφορες χώρες. Εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε τη φωνή των τοπικών μας συνομιλητών. Και ξέρω ότι οι αντιπροσωπείες της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, κάνει μια προσπάθεια βελτίωση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία διαβούλευσης. Όπως σας είπα και προηγουμένως, εμείς ακούμε πράγματα από τους ε, συνομιλητές μας, τους τοπικούς συνομιλητές μας. Και καμιά φορά η εικόνα που προκύπτει είναι μεικτή. Όταν παίρνουν ε, κονδύλια οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, υπάρχει μια καλή επικοινωνία αλλά συχνά υπάρχουν οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για την κοινωνία των πολιτών σε δύσκολες ε, συνθήκες, σε δύσκολες χώρες. Συχνά δεν μπορεί να επιβιώσει. Δεν έχει πρόσβαση, ας πούμε, στο ίντερνετ. Δεν έχει πόρους για να επιβιώσει, για να επιβιώσουν οι οργανώσεις της. Εμείς επίσης πιστεύουμε ότι η αποκέντρωση, κάτι που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και αυτό το χρηματοδοτικό μέσο ε, προωθεί την ε, επιτόπια διαχείριση των προγραμμάτων. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλό να γίνει συστηματικά μια διαβούλευση με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών επιτόπου δεν νομίζω ότι είναι θέμα θέλησης, ότι λείπει η θέληση. Συχνά οι αντιπροσωπείες ε, της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν τους πόρους για να κάνουν κάτι τέτοιο. Ακριβώς γι' αυτό πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Μια και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ε, έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία, όλος αυτός ο διάλογος. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικοινωνήσει και να συνδιαλλαγεί με την κοινωνία των πολιτών η Ευρωπαϊκή Ένωση. για τους στόχους ε, του χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το χρηματοδοτικό μέσο είναι καταπληκτικό ένα μέσο το οποίο προσπαθεί να βοηθήσει απευθεία τις οργανώσεις ε, τη κοινωνία των πολιτών, χωρί να περνάει μέσα από την και να προποθέτει τη συνένεση των ε, κυβερνήσεων. Αυτή η ικανότητα να παρακάμπτουμε την συνένεση των ε, κυβερνήσεων των τρίτων χωρών είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί έτσι εστιάζουμε στις πραγματικές ανάγκες των οργανώσεων της ε, κοινωνία των πολιτών. Γιατί πραγματικά θα θέλαμε, έτσι λοιπόν θα θέλαμε αυτό το μέσο να πρικοδοτηθεί με περισσότερα κονδύλια. Ούτω ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες, στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε προηγουμένως, ότι η Κομισιόν δηλαδή δεν θα εκπληρώνει διάφορες προϋποθέσεις, ας πούμε, της προβλεψιμότητας, λόγω έλλειψης πόρων, λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού. Επίσης, υπάρχει και μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος που ακυρώθηκε γιατί δεν είχαμε αρκετά λεφτά. Αυτά τα πράγματα με περισσότερα κονδύλια δεν θα συμβαίνουν. Το μέσο αυτό πραγματικά είναι απαραίτητο, αλλά για να υλοποιήσει το στόχο του θέλει περισσότερα λεφτά. Ανάλογα με τους στόχους που προωθεί. Επίσης, ε, οι στόχοι θα πρέπει να γίνουν πιο φιλόδοξοι ε, σε γεωγραφικό και θεματικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις απόψεις που μας εκφράσατε. και οι δύο τονίσατε τη σημασία της διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς. Τονίσατε επίσης το θέμα του προϋπολογισμού του χρηματοδοτικού μέσου. Θα πρέπει ο προϋπολογισμός να είναι στο ύψος των προσδοκιών. Και επίσης είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ε, κεντρομόλα τάση όλων των σχετικών εργαλείων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους διάφορους βουλευτές. Μία σειρά από βουλευτές. Η κυρία Λόχ Μπίλερ ούτω ή άλλω είναι υπεύθυνη εξ των Πρασίνων για την ε, αλλαγή του σχετικού κανονισμού. Νομίζω ότι ο, ο καθήλυνα αρμόδιο εισηγητή θα είναι από το ΕΛΚ, αλλά νομίζω δεν έχει ήδη προσδιοριστεί. Ξεκινάμε πάντως με την κυρία Γκόμε. πρώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, όπως το είπε ο κύριος Τίμας, ότι αυτό το μέσο τρέχει πάρα πολύ λίγο χρόνο. Παρ' όλα αυτά όμως, μπορούμε να επισημάνουμε κάποια προβλήματα που έχει. Άρα είναι σωστό να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε τα κακοσκήμενα τώρα στην ενδιάμεση φάση στην οποία βρισκόμαστε. Μπράβο, Πρόεδρε, που φωνάξατε τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική, ούτως ώστε να έχει νόημα η προσπάθειά μας. Θυμώ πάρα πολύ την σοβαρή συνεισφορά τους. Επίσης θα πρέπει να σας πω από προσωπική εμπειρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και από την εμπειρία μου στην Επιτροπή Ανάπτυξη ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω με τόσο μαζί είπαν οι ΜΚΟ. Διαβούλευση στη βάση από τις αντιπροσωπείες και το οποίο τώρα πάσχει. Και αυτό είναι σημαντικό και, με, και για το μέσο συνεργασία που έχουμε αλλά και για την υπαδιαρμοστία. Για το χρηματοδοτικό μέσο από την άλλη μεριά. Άρα θα πρέπει να φροντίσουμε οι αντιπροσωπείες μας επί τόπου να κάνουν ό,τι χρειάζεται τόσο ώστε να μπορούμε να, να ε, ε, αξιοποιήσουμε και το χρηματοδοτικό μέσο το ένα και το άλλο. Επίσης, θα πρέπει και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα πρέπει να ενταχθεί στις ε, θεματικές προτεραιότητες. Επίσης, η διαθέσιμη πόρη είναι περιορισμένη. Και στην πραγματικότητα η πρικοδότηση είναι μικρή διότι η Μύρδα του λέοντος πηγαίνει στις ε, αποστολές των παρατηρητών εκλογών. Έχουμε μια ομάδα εργασία που ασχολείται με αυτά, οπότε θα πρέπει να συνοδούμε και με αυτού. Γιατί θα πρέπει να αξιοποιούνται οι πόροι. Και όπως τα είπε και η εκπρόσωπος του δικτύου, θα πρέπει κάποια αλλαγή στον προπολογισμό να μπουν στα γεωγραφικά προγράμματα οι αποστολές ε, των, των εκλογικών παρατηρητών. Όμως η δική μου εμπειρία λέει ότι θα πρέπει να συνεχίσει να είναι αρμόδια η διεύθυνση της ΡΕΛΕΚΣ αλλιώς θα απονευρωθεί όλη η υπόθεση. Θα έχουμε ακόμα ένα χρηματοδοτικό μέσο για να ευχαριστήσουμε κάποιες κυβερνήσεις. Μπάσκετ προχωρήσουν περισσότερο στον εκδημοκρατισμό. Επομένως, να συνεχίσει και αυτό το πρόγραμμα Όμω, Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πόροι αξιοποιούνται και ότι πολύ περισσότερα χρήματα πηγαίνουν σε κάποιες δράσεις που πρέπει να πάνε. πρόληψη κρίσεων, ειρήνευση, εμπλοκή κοινωνίας των πολιτών. Τα θέματα καταπολέμησης βίας κατά γυναικών και ανηλίκων, καταπολέμηση δυσμενών διακρίσεων και τις άλλες υποστηρικτικές δράσεις που έχουμε για βασανισμούς, ανήλικους στρατιώτες, πιθανωτική ποινή και βία κατά γυναικών και ανηλίκων. Basically... Αυτά ήθελα να πω βασικά. Επίσης επαναλαμβάνω ότι συμφωνώ με τον προβληματισμό τους ότι διαμορφώνεται μία τάση στην Επιτροπή μας να επιδιώκουμε οι πόροι να πηγαίνουν σε κάποιες δράσεις που είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο των κυβερνήσεων. Πρόκειται για ένα μέσο πάρα πολύ σημαντικό. Άρα να πηγαίνει σε κάποια προγράμματα που, είναι, που δεν συνδέονται, δεν, δεν χρειάζονται συνένεση, σύμπραξη των κυβερνήσεων. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Σήμερα το πρωί πρέπει να σας πω η, η Κομισιόν συμμετέσχε σε κάποιο συμπόσιο, μια εκδήλωση για τα δικαιώματα τη γυναίκα και για το πρόβλημα τη βία. Επισημάνθηκε πρόβλημα με τον προπολογισμό, πρόβλημα ψυχοπρικοδότηση και άρα το θέμα είναι να δοθεί προτεραιότητα στα θέματα αυτά που μα ενδιαφέρει. Όπω τα θέματα υγεία, τα θέματα αντιμετώπιση τη βία. Να έχουν προτεραιότητα και έτσι να μην έχουν πρόβλημα χρηματοδότηση. Αντρικέν. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα, γνωρίζουμε ότι ο στόχος 1 στα έγγραφά μας λέει ότι εφαρμόζεται σε χώρες όπου διαπιστώνονται συστηματικές και συνεχείς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από κάτω γράφει για παράδειγμα ε, ε, περιορισμό της ανεξιθρησκείας. Μιλήσαμε και με μια αντιπροσωπεία ε, από τις Ηνωμένες που μιλήσανε για freedom of religion. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να ε, χρηματοδοτήσει προσπάθειες για το θέμα αυτό από τον προπολογισμό αυτό και ποια ήταν η προηγούμενη πρακτική από το 2007 σχετικά με την χρηματοδοτική υποστήριξη τέτοιων ε, σχέδιων. Και δεύτερο σύντομο ερώτημα. Ποια είναι η στρατηγική της Κομισιόν για την υποστήριξη δράσεων που καλύπτονται από ευρωπαϊκές κατευθυντήρες γραμμές ιδίω για ανθρώπινα δικαιώματα, διάλογο και διαβουλεύσεις με χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν, όπου ο διάλογος αυτός δεν καταλήγει ε, σε πλήρωση των στόχων σύμφωνα με τις προσδοκίες μας. Θα περιληφθεί στη νέα στρατηγική σας 2011-2013. Κίτος λέει πρόεδρος. Κυρία Ντεκάιζερ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ για να καταφέρουμε να υλοποιηθεί αυτό το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ήταν καθόλου κάτι το δεδομένο. Και ο περιορισμένος προϋπολογισμός του προφανώς δεν μας ικανοποιεί. Καταλαβαίνω βεβαίω την απογοήτευση, ειδικά των μη κυβερνητικών οργανώσεων, για το γεγονό αυτό. Το ερώτημά μου αφορά την αξιολόγηση. Η Κομισιόν μας λέει ότι πρόκειται για ένα νέο μέσο που είναι σε μια φάση εξέλιξης και ανάπτυξης και ότι δεν είναι ακόμα δυνατό σήμερα να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα και κάποια διδάγματα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής στην Κομισιόν. Έμαθε τίποτα από την έκθεση που έγινε πέρυσι στην προηγούμενη κοινοβουλευτική ε, θητεία και την ε, συντάξαμε εγώ και μια συνάδελφος όπου καναμε μια αξιολόγηση των εκλογικών αντιπροσωπιών που χρηματοδοτούνται από αυτό το μέσο. Ε, τονίσαμε ότι υπάρχουν δυσκολίες με τη χρηματοδότηση αυτών των αποστολών, ότι είναι σημαντικές οι αποστολές αυτές, ε, ότι υπάρχουν διάφορα κενά που θέλουμε να καλυφθούν και αυτό που μα ενδιαφέρει είναι και τι γίνεται μετά τι εκλογέ, τι follow-up υπάρχει, τι συνέχεια δίνεται. Η Κομισιόν έκανε κάτι με την εκθεσή μα, σκοπεύει να κάνει κάτι με την εκθεσή μα. Γιατί όχι απλώ ανασκουμποθήκαμε και δουλέψαμε πολύ για αυτή την έκθεση, αλλά πληρώσαμε και έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα στην ΑΦΕΤ για να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση. Θα ήταν κρίμα σήμερα να μην μάθουμε τίποτα από αυτή την έκθεση. Έτσι, μια ερώτηση προς την Κομισιόν και θα ήθελα να μου απαντήσει. Ευχαριστώ. Κυρία Ντεκάιζερ. Κύριος Χόβιτ. Ευχαριστώ. Πραγματικά ε, δυσαρεστήθηκα για το γεγονός ότι άλλαξε η ημερήσια διάταξη από τη μία, αλλά από την άλλη είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Είναι χρήσιμο να συζητήσουμε και με τους ε, εκπροσώπους της Κομισιόν πριν υποβάλουν το έγγραφό τους. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Τίμα στην αρχή, ότι ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές, όσοι περίμεναν ουσιαστικές ή ριζικές αλλαγές, ε, ας, είναι πιο ρεαλιστές. Εγώ ούτως ή άλλως ήμουν υπεύθυνη για τις αρχικές ε, τροπολογίες και θέλω να δω με ενδιαφέρει να δω τι εξέλιξη θα ακολουθήσει. Και θα παρακολουθήσω και τις εξέλιξεις στον κανονισμό. Όταν μιλάμε για τις ε, προτεραιότητες που δίνουμε, για το ΦΠΑ, για το, τη σχέση με το DCI, Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι, σχετίζονται κιόλα με την αποτελεσματικότητα του προϋπολογισμού. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό το μέσο είναι το βασικό μας μέσο που έχουμε για να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο ε, και τη δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι συζητήσεις. Καλό είναι λοιπόν να μην τις ε, πνίξουμε μέσα στις δικές μας εσωτερικές ας πούμε, συζητήσεις, στην ε, δική μας κουζίνα και στα δικά μας μαγειρέματα. Κοιτάξτε, δεν περιμένω πλήρης απαντή σήμερα το πρωί. Θα ήθελα όμως να δούμε κάποια από τα δύσκολα θέματα του και πού συμφωνούμε για τον κανονισμό. Καλό θα είναι να δούμε τι έχει γίνει για αυτά τα πράγματα. Ε, επίσης όλα αυτά τα θέματα δεν τα έχουν φύξει όλα ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Καταρχάς το θέμα του ρίσκου. Ε, συχνά μας κατηγορούν ότι το παίζουμε, ότι κινούμαστε εκ του ασφαλού. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ με αυτό το μέσο είναι πραγματικά καινοτόμο και επικίνδυνο. Ε, το θέμα του πόσο μπορούμε να συνεργαστούμε με τα κομμάτια της αντιπολίτευσης, ας πούμε. Ε, γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν φεζόνες ανάμεσα στη σχέση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το θέμα είναι πόσα ρίσκα έχουμε πάρει και πόσο έτοιμοι είμαστε να αποτύχουμε. Δεύτερον, το θέμα του mainstreaming. Αναφέρθηκε από τις συναδέλφους. Εμείς είχαμε πει ότι θέλουμε ένα ξεχωριστό μέσο, αλλά δεν θέλουμε να έχει αρνητικές επιπτώσεις αυτό που γίνεται ε, με τα γεωγραφικά προγράμματα, που είναι οι βασικές μας πολιτικές. Θέλουμε να αλληλεπιδρούν αυτά τα δύο μέσα για να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα να ακούσω τι λέει ο αξιολογητής ε, για αυτό το θέμα. Είμαι πεπισμένος ότι πράξαμε το σωστό, αλλά τα πράγματα στην πράξη πώς ε, υλοποιήθηκαν, πώς εξελίχθηκαν. Ε, έχω δίκιο με αυτά που λέω. Επίσης, το ίδιο με αυτό που είπε η συνάδελφος για τις ε, αποστολές παρατήρησης εκλογών. Είμαστε περήφανοι για αυτές τις αποστολές και δεν θέλουμε να τις περικόψουμε. Το πρόβλημα με το μέσο είναι τα χρήματα, γιατί οι αποστολές αυτές είναι πάρα πολύ ακριβέ και είναι ακριβέ γιατί τι κάνουμε καλά. Να το πούμε τίμη, έτσι. Ε, θα μπορούσαμε να ξοδέψουμε και ακόμη περισσότερα για τι αποστολέ αυτέ και θα ήταν και δικαιολογημένο. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα ε, σε αυτό, να το κάνουμε καλά, τι αποστολέ αυτέ, αλλά να μην γίνεται ει βάρο τη υπεράσπιση των α, ε, α, ε, ακτιβιστών των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Το θέμα δεν είναι ότι θέλουμε περισσότερα λεφτά. Πάντα θέλουμε περισσότερα λεφτά. Το θέμα είναι ε, να προωθήσουμε παράλληλα και τους δύο στόχους μέσα στην πρωτοβουλία αυτή, μέσα στα πλαίσια του χρηματοδοτικού μέσου. Και τέλος, πόσο επιτακτικοί είμαστε, πόσο, πόσες ε, υποδείξεις βάζουμε. Ε, πρέπει να το κάνουμε αυτό ή θα πρέπει να είμαστε αρκετά ανοιχτοί και αρκετά ευέλικτοι. Ε, όταν υπάρχουν ανάγκες, όταν συμβαίνει μια κρίση, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι και ούτε πρέπει να επικρίνουμε την ε, Κομισιόν. Αλλά αυτά είναι βασικά θέματα και ελπίζω τουλάχιστον, τουλάχιστον να τα θέσουμε ε, και να, είναι, να αποτελέσουν τμήμα μιας μελλοντικής συζήτησης. Σας ευχαριστώ κύριε Χάριτ. Κύριε Λορμπιλέ, παρα, παρακαλώ ωστόσο όλες και όλοι να είστε σύντομες και σύντομοι για να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Κύριε Λόρμπιλερ, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ που είμαι και νέα Ευρωβουλευτής τα βρίσκω πολύ εντυπωσιακά το τι έχει γίνει δηλαδή με τα χρήματα αυτά και τη χρηματοδότηση αυτή. Ε, τα βρίσκω καλά. Ακούω όμως ότι πολλά καλά project απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Λέω λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι πολύ υψηλότερος και ίσως μάλιστα πρέπει να εξετάσουμε και το ερώτημα ποια project θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τούτο εδώ το μηχανισμό και ποια από άλλα, όπως για παράδειγμα προενταξιακά. Στη συζήτηση λοιπόν που θα κάνουμε περαιτέρω Νομίζω ότι αυτό ίσως είναι ένας τρόπος να εξασφαλίσουμε περισσότερα χρήματα για ε, έργα, project ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως είπατε, η επίτροπο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα πέρασε από εδώ και είπα ε, ότι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τα χρήματα αυτά. Είπε όμως ότι και οι ανάγκες ε, ε, έχουν αυξηθεί και ζήτησε περισσότερη χρηματοδότηση. Όπως είπαν άλλωστε οι εκπρόσωποι των μη κρατικών οργανώσεων, φαίνεται ότι υπάρχει ε, ανάγκη ενίσχυσης των αντιπροσωπιών της Ένωσης στις διάφορες χώρες επιτόπου για να ενισχυθεί και η συνεργασία τους και η διαδικασία να γίνει πιο να μπορέσει να συμπεριλάβει περισσότερους και να απλωθεί περισσότερο. Φαίνεται πως είναι μέχρι τώρα ε, λίγο ικανοποιητική η διαδικασία αυτή. Επίσης επιθυμώ να υποστηρίξω τα όσα είπε ο κύριος Τίμανς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σωστό να περιληφθούν και τα οικονομικά, κοινωνικά δικαιώματα γιατί ε, είναι σημαντικό να ενισχυθούν τα συνδικάτα, να καταπολεμηθεί η εξαναγκαστική εργασία είναι λοιπόν το ίδιο σημαντικά και τα συλλογικά δικαιώματα. Άκουσα ότι έχουν ληφθεί και αποφάσεις στο παρελθόν που αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν ορθές. Για παράδειγμα, η απόφαση που έχει ληφθεί δεν ε, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν ε, θεραπευτικά κέντρα για όσους έχουν υποστεί ε, ψυχολογικούς, ψυχολογικούς τραυματισμούς από ε, βασανιστήρια. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για λογαριασμό της χώρας μου, της Γερμανίας. Η χρηματοδότηση τριών μόνο κέντρων, λέει η χώρα μου, είναι επαρκής. Αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Υπάρχουν λοιπόν και μεμονωμένε αποφάσει οι οποίε δεν έχουν βελτιώσει την ατζέντα των ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά έχουν μάλλον ε, οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. Και τέλος η ερώτησή μου, διάβασα ότι δαπανάτε πολλή ενέργεια για περισσότερη ορατότητα και καλύτερη επικοινωνία για το μηχανισμό αυτό. Και αυτά θεωρώ ότι είναι καλά πράγματα. Αλλά αξιολογούμε επίσης εάν αυτά είναι επαρκή. Εάν για παράδειγμα υπάρχει μια λίστα διασταυρούμενων θεμάτων χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο τα διαθέσιμα χρήματα ώστε να μπορούν να γίνουν ε, να γίνει επικοινωνία για τα θέματα αυτά. Γκέρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με αυτό το τελέξαν για τα κενά του προβολισμού που είναι κάτι το απαράδεκτο νομίζω ότι θα πρέπει να διορθώσουμε την ανεπάρκεια των πόρων όσο είναι δυνατό. Υπάρχουν τώρα και κάποια άλλα ε, προβλήματα ε, εγγενή στο σύστημα ε, λήψης απόφαση όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά εμπόδια έχουμε. Η Real Politik πρώτα-πρώτα που είναι σαν σταυρός Μα με 150 χρόνια τόσο να μπορούσαμε να κωδικοποιήσουμε τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Οπότε τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να πέρασαν 150 χρόνια μέχρι και να κάνει κάτι αντίστοιχο για να τα κατοχυρώσει. Να συμφωνήσουμε επομένω ότι κάτι πρέπει να γίνει για αυτά τα βασικά θέματα. Αλλά να συμφωνήσουμε κατά πόσο το δικαίωμα στη διατροφή είναι, είναι δικαίωμα ε, του ανθρώπου, είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Οπότε και έτσι θα μπορούμε να δούμε κατά πόσον αυτό το δικαίωμα υπάγεται ή όχι στα θέματα γεωστατικής πολιτικής. Η οχι στα θεματα γεωστατικης πολιτικης η Να μας πει η Κομισιόν πώς βλέπει αυτό το, το, το, το, ερώτημα. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα στον τογετό. Είδατε πόσοι φραγμοί, πόσοι εμπόδια υπάρχουν γι' αυτό σε όλο τον κόσμο. Το δικαίωμα διατροφής επομένως. Τι είναι, είναι κάτι που αναφέρεται στα εγχειρίδια βιολογίας είναι δικαίωμα του φυσικού προσώπου. Το δικαίωμα στον εμβολιασμό, τι είναι, είναι δικαίωμα. Δηλαδή το, το επιφυλάσσουμε για το ένα δισεκατομμύριο δικούς μας και, άλλα και, και τα άλλα πέντε δισεκατομμύρια τίποτα. Οπότε αυτοί δίνουν τα λεφτά και βολεύονται μόνο οι πλούσιοι. Αυτό σας λέω. Να κάτσουμε και να σκεφτούμε και να διερευνήσετε με τους συνεργάτες σας σε συνεργασία και με δύο-τρεις βουλευτές και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρόκειται για οριζόντιο θέμα να δούμε τα εμπόδια που υπάρχουν στι διεθνεί διαπραγματεύσει, κυρίω στον ΠΟΕ. Πώ θα να με όλους τους εταίρους μας και κυρίως με την Κίνα. Και άρα με κάποιο έξυπνο τρόπο να βρω μια λύση. Κάντε επομένω ε, μια, μια τέτοια διερευνητική ομάδα. έτσι άτυπα. Ούτως ώστε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να κωδικοποιήσουμε αυτά τα δικαιώματα, τα οικονομικά και κοινωνικά. Μου φαίνεται πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Να δούμε επίσης και ποια είναι η πιο δόκιμη στρατηγική για να σημειώσουμε κάποιο πρόοδο. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκέρεντς για τις παρατηρήσεις σας που ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες. Κυρία Όιλαντ αρχίζει να μας πιέζει και ο χρόνος πια. Ζητώ συγγνώμη, πάντα οι τελευταίοι την πληρώνουν, οι τελευταίοι ομιλητές έχουν λιγότερο χρόνο, αλλά τι να κάνουμε, έτσι γίνεται. Γιατί θα ήθελα να δώσω και το λόγο και στην ε, Κομισιόν και στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Έχουμε και έναν προσκεκλημένο από την ε, Νιγηρία. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Ευχαριστώ. Το θέμα που θέλω να θέσω απαιτεί περισσότερο χρόνο. Είμαι νέο μέλος και στο Κοινοβούλιο και στην Υποεπιτροπή και συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπατε. Η ατζέντα αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα σας πω κάτι που δεν πρέπει να το πάρετε στραβά. Νομίζω όμως ότι το θέμα αυτό το σημερινό θυμίζει το χθεσινό, θυμίζει το παρελθόν δηλαδή. Ε, πρέπει να δούμε, ε, να στραφούμε προς το μέλλον πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις υπανάπτυκτες χώρες να αλλάξουν την κοινωνία τους, να εκδημοκρατιστούν, να ανοίξουν, να είναι κοινωνίες που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που εννοώ ε, είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα ε, να επενδύσουμε ε, στην κοινωνία των, ε, της τεχνολογίας, στα σχολεία. Οι, οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να μπουν στα σχολεία. Θα πρέπει οι νέες γενιές να μάθουν τους υπολογιστές, να μην είναι αναλφάβητες ψηφιακά. Ε, στις σημερινές κοινωνίες υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και η πρόσβαση στην ελεύθερη ενημέρωση είναι βασικό δικαίωμα. Ζούμε στον 20ο αιώνα στο κάτω, πρώτο αιώνα στο κάτω-κάτω. Και η ενημέρωση και οι τεχνολογίες ενημέρωσης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αν επενδύσουμε σε αυτές τις χώρες, σε αυτούς τους τομείς, νομίζω ότι επενδύουμε πραγματικά στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μπουράτσης, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός, γιατί ακούστηκαν πολλά και προτάθηκαν πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσω και εγώ λοιπόν να είμαι συνοπτικός και να αναφερθώ σε συγκεκριμένα γεγονότα και στοιχεία. Ξεκινάω από ένα θέμα που το έθιξε και η εκπρόσωπος ε, του Concord και η κυρία Γκόμες. Δηλαδή, κάτι που αφορά την άμεση χρηματοδοτική υποστήριξη. Και θέλουμε άμεση χρηματοδοτική υποστήριξη ή θέλουμε να δίνουμε τα χρήματα πρώτα στις ΜΚΟ. Σε όλες τις ε, προσπάθειες αναπτυξιακής βοήθειας ε, η τάση ε, να τη χρηματοδοτούμε είναι με ένα ποσοστό 25%. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεύτερο στοιχείο. Φέτος, το 2009, θα ξοδέψουμε για τις ε, εκλογές 23 εκατομμύρια, όχι παραπάνω. Άντε, 23-24 από τα 140 εκατομμύρια. Επομένω, τη μερίδα του λέοντο δεν την παίρνουν οι αποστολέ παρατήρηση εκλογών. Ένα τμήμα πηγαίνει εκεί, αλλά σίγουρα όχι η μερίδα του λέοντο. Πρέπει να τα διευκρινίσω αυτά. Ζητώ συγγνώμη. Προσπαθούμε να κάνουμε οικονομίες, ούτω ώστε να βοηθήσουμε και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Λοιπόν, τι είναι μύθος και τι είναι πραγματικότητα στη διαβούλευση. Αυτό συνδέεται επίσης και με το θέμα που τέθηκε από την κυρία Μπίλερ. Για τα λεγόμενα προϊόντα επικοινωνίας, τα επικοινωνιακά προϊόντα. Διαβούλευση. Πριν από την αποκέντρωση, πριν το 2003-2004, οι αντιπροσωπείες μας δεν ασχολούνται με τέτοιου τύπου ερωτήματα. Ειδικά μάλιστα στον τομέα ειδικά στο θέμα της, των σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών. Από το 2003-2004 για την προσωπίες μας έχουν περισσότερη δουλειά. Βεβαίως έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά δεν είμαστε ακόμα τέλειοι. Και για να σας δείξω ότι υπάρχει πρόοδος στην ε, διαβούλευση, ε, σας παραπέμπω στην έκθεση του Concord. Κάθε χρόνο συντάσσεται για, την, ε, για τις εξελίξεις της διαβούλευσης. Και η έκθεση λέει ότι η διαβούλευση βελτιώθηκε σαφώς τα τελευταία χρόνια. Κάτι το οποίο είναι προφανές από τη στιγμή που έγινε αποκέντρωση. Δεύτερη απόδειξη για του λόγου μου, του λόγου μου το αληθές. Είναι το ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο μίλησε και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, στην Επιτροπή Ανάπτυξης και στο για το Συμβούλιο και είπε ότι όντως υπάρχει βελτίωση στη διαβούλευση των αντιπροσωπιών. Ε, μερικές φορές βέβαια οι αντιπροσωπείες μας ερμηνεύουν διαφορετικά τις οδηγίες μας. Υπάρχει διαφορετική ερμηνεία. Αλλά βέβαια οι ερμηνείες αυτές δεν θα πρέπει να διαφέρουν τόσο πολύ. Θα έπρεπε δηλαδή να, να ακολουθούν όλες οι αντιπροσωπείες το ίδιο εγχειρίδιο, για να το πω έτσι. Σε ό,τι αφορά τα επικοινωνιακά ε, προϊόντα, τα λεγόμενα. Ε, κάνουμε ενημέρωση για τα βασανιστήρια και για άλλα θέματα ε, μέσω συνεδριάσεων που, κάνουν, που οργανώνουν οι διάφορες αντιπροσωπείες και μέσω ε, διαφόρων προβολών, ας πούμε. σε καμία περίπτωση, ό,τι και να κάναμε, ό,τι και να προβάλαμε εμεί τι δικέ μα οθόνε, καμία κρατική τηλεόραση δεν μπόρεσε ποτέ δεν πήρε ποτέ ας πούμε, αυτά τα προϊόντα τα δικά μας ας πούμε, για να τα μεταδώσει εθνικά. Το, ο μόνος, η μόνη τηλεόραση ε, ή τα μόνα μέσα που αγοράζουν το εισαγωγικών τα προϊόντα μας είναι ο ΙΕ. Κυρία Γκόμες, ελπίζω να είστε στο Χόλμη την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να σας πω το εξής. Εμείς έχουμε θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, στο επίκεντρο του European Development Days, ε, του γεγονότος αυτού, της εκδήλωσης αυτής που θα γίνει στη Στοκχόλμη. Ένα μεγάλο, μια μεγάλη εκδήλωση που οργανώνει η Σουηδική Προεδρία. Κέντρα αποκατάσταση τώρα. Όλοι, όλοι λοιπόν γιατί είναι δεδομένη η απόφαση του Συμβουλίου, τόσο ώστε να υπάρξει αυτή η μεταβολή από το χρόνο να, να υπάρχει θυλαγή όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ταμεία. Όμως έχουμε τα υπάρχοντα τα οποία σας παρακαλώ λέει ο Πρόεδρος αν μπορείτε συνοψίστε τελειώνω τελειώνω κυρία Merci. Yeah, Mr. Timas, but as, as you both know, we have the working group on the institute. Έχουμε μια ομάδα εργασίας για το μηχανισμό αυτό, άρα δηλαδή θα μπορέσουν τα μέλη μας να εγκύψουν στις λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να το πράξουμε τώρα εδώ. Κύριε Τίμαρς, εσείς για τη στρατηγική. Εγώ βρήκα ε, την συζήτηση και τις ερωτήσεις των αξιοτήμων ευρωβουλευτών ενδιαφέρουσες. και πολλές από αυτές αξίζουν να συζητηθούν σε μεγαλύτερο βάθος. Όμως, όπως τα γνωρίζει η γραμματεία της υποεπιτροπής σας, έχω ζητήσει από καιρό, από πολλές εβδομάδες, ε, ε, ανεπίσημη συνεδρίαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα του Μηχανισμού Διαβουλεύσεων και Στρατηγικής δεν θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Θα έρθω σε λίγα θέματα μόνο. Εμεί οι ίδιοι πρώτοι λέμε βεβαίω αν μπορεί να μα δοθεί μεγαλύτερο προπολογισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μακάρι δώστε μα, Αλλά δεν περνάει από τα δικά μα χέρια. Σε ό,τι αφορά τη διαβούλευση στο τοπικό επίπεδο θα κάνουμε προσπάθεια μαζί με του ε, συναδέλφου μα να ζητήσουμε από τις αντιπροσωπείε μα να εγκύψουν περισσότερο στο θέμα. Μη λησμονείτε ωστόσο ότι οι αντιπροσωπείες μας ε, βρίσκονται εν ώψη μεγάλης αναστάτωσης όταν θα ε, τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της ε, Λισαβόνας και θα χρειαστεί βεβαίως να εξορροπηθούν με προσοχή οι προτεραιότητες. Για την κυρία Γκόμες, ο ICC είναι ήδη βασικός στόχος χρηματοδότησης του στόχου 4 δηλαδή η βία κατά, τη, κατά των γυναικών και των νέων κοριτσιών περιλαμβάνεται ήδη στη στρατηγική μας η καταπολέμησή της δηλαδή και θα περιληφθεί και στις νέες κατευθύνσεις γραμμές για την κυρία Αντρικιένε η θρησκεία, η ελευθερία δηλαδή άσκησης της θρησκείας είναι και αυτή μέσα στους στόχους Τη παρούση στρατηγική και θα διατηρηθεί. Και το θέμα το θέτουμε όχι μόνο μέσω του EIDHR αλλά και μέσα από όλο το φάσμα των προσπαθειών μας σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές κατευθυντήρες γραμμές για την διαβούλευση και τον διάλογο εμείς χρηματοδοτούμε μόνο τα σεμινάρια. Ο ίδιος ο διάλογος χρηματοδοτείται από τον επιχειρησιακό προπολογισμό της Κομισιόν. Γιατί την Κάιζερ Τεκάιζερ, σχετικά με την ε, ενδιαφέρουσα ερώτησή σας σχετικά με την συνέχεια που δόθηκε στην έκθεση τη δική σας και του κ. Σαλαφάνκα, ομολογώ ότι λησμόνησα να πω ότι υπό τον στόχο 5 και υπό τον στόχο 2 της επανεξέτασης θα κάνουμε ειδική αναφορά στην αναγκαία συνέχεια, follow-up, που πρέπει να δοθεί μαζί με την κοινωνία των πολιτών στις συστάσεις των παρατηρητών εκλογών. Αυτό προβλέπεται ρητά. Λυπούμε, ε, ε, διότι το ξέχασα να το αναπαντήσω προηγουμένως, βέβαια και άλλες συστάσεις ε, θα ληφθούν υπόψη. Ο Χάουιτ έθεσε ορισμένα σημαντικά θέματα που δεν νομίζω ότι μπορώ να συζητήσω τώρα μαζί του, άλλωστε έχει, είναι απόν πλέον. Ε, θα μου μείνει η κυρία Λόχμπίλερ τώρα, αύξηση του προϋπολογισμού, η υποστήριξη του γραφείου του ύπατου εκπροσώπου εγγράφεται μέσα στις υποχρέσεις του HDR. Είναι η μόνη διεθνής οργάνωση που λαμβάνει χρηματοδότηση διαρκή που δεν είναι, έχει γίνει air marked από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η χρηματοδότηση που λαμβάνει το γραφείο είναι περίπου τη ύψη των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Είχαμε φροντίσει τότε να εγγραφεί αυτό στο κείμενο του κανονισμού. Σχετικά με την πρόταση του κ. Γκέρενς, δεν μπορώ να του υποσχεθώ αυτή τη στιγμή ότι θα δημιουργηθεί ένα μια τέτοια ομάδα, ένα τέτοιο κύτταρο διερεύνησης. Είναι κάτι που πρέπει ίσως να συζητήσει η Επιτροπή Ανάπτυξης και η δική σας υποεπιτροπή. Ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρόκειται να παραμείνει κλειστή απέναντι σε αυτή τη συζήτηση. Υπενθυμίζω, ας κάνουμε την ε, ομάδα εργασίας όσο γίνεται νωρίτερα και μπορούμε να προχωρήσουμε τότε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ασφαλώς την πρόθεση να οργανώσουμε την συνάντηση αυτή το δυνατόν συντομότερο, διότι πρόκειται η προτεραιότητα και δική σας και δική μας, της Υποεπιτροπής δηλαδή. Θα γίνει επομένω αυτή η συνάντηση, σας βεβαιώ. Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι οι βουλευτές μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία για να ζητήσουν συμβουλές όταν συμμετέχουν σε αντιπροσωπείες επιτόπου. Ιδίω όταν πρόκειται για χώρες που έχουν ενδιαφέρον για τον HTCI μπορείτε να ρωτήσετε για παράδειγμα όταν μεταβαίνετε στη Τουρκία να μάθετε ποιοι είναι οι μηχανισμοί που χρηματοδοτούνται από αυτό. Ε, Ποιε είναι οι οργανώσει, οι τουρκικέ οργανώσει οι οποίε χρηματοδοτούνται και ούτω καθεξής. Θα τα πούμε όμω αυτά την επόμενη φορά. Σα υπενθυμίζω ότι έχουμε την προφορική ερώτηση την τρίτη από ό,τι φαίνεται τη επόμενη εβδομάδα. Εξάλλου. Δεν υπάρχει συνέχεια σε την, δεν έχει συνέχεια σε αυτή την αίτηση που είχε γίνει από πλευρά ε, της Επιτροπής. Τώρα, ε, στο 6 έχουμε ένα θέμα. Βουλευτές διεθνούς δράσης. Έχουμε κοντά μας ένα γερουσιαστή από την Ιγυρία. Σήμερα γίνεται μια συζήτηση η οποία διεξάγεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διεθνή θέματα. Και γι' αυτό θελήσαμε να περιλάβουμε το θέμα αυτό. Καλώ ήρθατε κύριε Γερουσιαστά. Ο κύριος Πρόντι, από όσο ξέρω, έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, Ένωσης Βουλευτών. Κύριε Πρώτη, μπορείτε εσείς να απευθύνετε λίγα λόγια στον ε, γερουσιαστή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί σε λίγο στο 5G2 2 εχω μια άλλη συνεδρίαση για μια άλλη πρωτοβουλία που αφορά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο όπου θα παραστεί και ένας δικαστής συγκεκριμένα ο πρόεδρος του δικαστηρίου ο κύριος Σούγκ είναι προσκεκριμένοι όλοι οι συνάδελφοι στο 5G2 2 θα γίνει αυτή η συνάντηση τόσο ώστε να μπορούμε να ενημερωθούμε όσον αφορά τώρα και αυτή την πρωτοβουλία Parliamentarians for Global Action. Πρόκειται για μια ε, ε, ένωση, για μια ομάδα ε, βουλευτών που προσπαθούν να εκπονήσουν μια στρατηγική ούτως ώστε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να κατοχυρωθεί σε σχέση με τη συνθήκη της Ρώμης. Στην, ε, στην ε, Ιαπωνία επίσης έχουν γίνει και προσπάθειες. Οι ΙΠΑ ακόμα δεν έχουν προσχωρήσει αυτό το, το σκοπό. Ε, γιατί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που θα πρέπει να επιληθούν ακόμα ισχύουν. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, λέει η Πρόεδρος. Καλώς ήρθατε και πάλι κύριε Γερουσιαστά. Δυστυχώς όμως έχουμε εξαντλήσει το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρουσα την συζήτηση, αλλά έχετε στη διάθεση σας τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Λέω Γιώργος Σωστής. Ναι, μεγάλη μου τιμή και ικανοποίηση να είμαι εδώ ε, όχι μόνο ως πρόεδρος αυτής της ε, Ένωσης Βουλευτών αλλά και ως πρόεδρος ε, Κοινοβουλίου της Νιγηρίας. Ε, έχω διατελέσει πρόεδρος σε αυτήν την Ένωση Βουλευτών τελευταία διετία. Το BGA είναι ένα δίκτυο βουλευτών. χίλιοι βουλευτές περίπου από 130 κοινοβούλια. Σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε διάφορα προγράμματα τα οποία επιμελούμεθα και η βιώσιμη ειρήνη και η δημοκρατία ε, είναι ένα πρόγραμμα είναι άλλο για το διεθνές δίκαιο και τη δημοκρατία είναι τα πιο προβλημένα μας ε, προγράμματα θέλουμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε το να προσχωρήσουν στην ε, Σύμβαση της Ρώμης, όλοι. Και 65, 65 ε, ε, χώρες καταφέραμε να προσπογράψουν την συνθήκη της Ρώμης. Άρα καταλαβαίνετε ότι δουλεύουμε σκληρά. Η Χιλή και η Τσέχη το 2009 είναι οι πιο πρόσφατες κατακτήσεις μας. Κουκ, νησιά Κουκ, Σουρινάμ και Μαδαγασκάρη το 2008 είναι οι αμέσως προηγούμενες χώρες. Ως Νιγηριανός επιτρέψτε να σας πω ότι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δημοκρατία είναι κάτι που πάρα πολύ μας ε, ενδιαφέρει. Αναπτύσσουμε ιδιαίτερη δραστηριότητα στην Δυτική Αφρική γιατί προσπαθούμε να ε, εξασφαλίσουμε ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή αυτή και νομίζω ότι διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο. Στην ε, Λιβερία υπήρξε ε, επίσης μια ευκαιρία πρωτοβουλίας μας και τελικά ο πρόεδρος της Λιβερίας οδηγήθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Έχουμε συμφωνία εταιρικής σχέσης με χώρες και φορείς από την Ευρώπη και συνεργασία. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό. Όπως δεν γνωρίζετε, πριν από λίγες εβδομάδες ξέσπασε κρίση στην Γουινέα. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε η ομαλότητα να πρετανεύσει και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την κοινότητα της έχει ήδη επιληφθεί. Αν δεν γνωρίζετε, κάποιοι προσεκλήθησαν σε ένα γήπεδο όπου πολλοί από αυτούς ε, σκοτώθηκαν με πυροβολισμούς. Οπότε ο φορέα των βουλευτών το οποίο προείσταμε ασχολείται με ανθρωπίνα δικαιώματα, με τη δημοκρατία. Ε, κινούμαστε δύο από δύο άξονε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να απαγορευτούν τα ελαφρά όπλα και δεύτερον θέλουμε να καλέσουμε όσο γίνεται περισσότερες χώρες να προσωπεύουν την της Ρώμης. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόντι για την πρόσκλησή του. Ε, όπως είπε, στο 5G2 μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Εκεί θα έρθει για να μας μιλήσει ο πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Σας ευχαριστώ κύριε Γερουσιαστά για τα λόγια σας. αν γνωρίζαμε ποια ε, ήταν η κατάσταση προηγουμένως, θα μπορούσαμε να είχαμε οργανωθεί καλύτερα. Δυστυχώ τη σχετική πληροφόρηση την λάβαμε αργά. Εν πάση περιπτώσει, ο, ο πρόεδρο του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου είναι εδώ όπως είπατε. Για μένα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμπειρία όταν διαπίστωσα ότι ο πρώην πρόεδρος της Λιβερίας ε, βρίσκεται τώρα ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού, Δικαστηρίου. Ήταν όπως είπα σημαντική εμπειρία για μένα. Έχουμε λοιπόν ε, την ε, ένοχτη ε, βουλευτών για παγκόσμια δράση. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, το θέμα της Γουινέας που αναφέρατε κύριε Γερουσίστα θα συζητηθεί την επόμενη πέμπτη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα θα το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ όλους και όλους για τη συμμετοχή σας στην συνεδρίαση.